παρεμβάσεις του ενό λεπτού. Δίνω καταρχήν το λόγο στην κυρία Κουλπέκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Την ε, παραμονή της πρωτοχρονία σε πολλές πόλεις της Γερμανίας, σε δημόσιους χώρους, περίπου 200 μετανάστες επιτεθήκανε σε πολίτες, κυρίως γυναίκες, τους ε, κλέψαν τα πορτοφόλια, τους ε, παρενοχλήσαν κτλ. Αυτό φαίνεται ότι ήταν μια οργανωμένη ε, ενέργεια. Για μέρε η αστυνομία και τα μέσα ενημέρωση προσπάθησαν να κουκουλώσουν το θέμα αυτό και να κρύψουν την ταυτότητα των ενόχων για αυτέ τι επιθέσει. Αυτό δεν είναι μια αποδεκτή όμω αντιμετώπιση στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε με τον τρόπο αυτό να προχωρήσουμε. Οι κανόνε μα ισχύουν για όλου. Το κράτο δικαίου θα πρέπει να καλύπτει όλε τι ευρωπαϊκέ αρχέ. Όταν μιλάμε για Ευρωπαίου ή για μετανάστε, δεν υπάρχει καμία διαφορά. Όταν δεν τηρούν την νομοθεσία, θα πρέπει να δεχτούν τι συνέπειε. Οι συνέπειε πρέπει να είναι σοβαρέ. Είναι η ευθύνη λοιπόν των δραστών που πρέπει να αναγνωριστεί και πρέπει να πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα και αν <clears throat> υπήρχαν τα σωστά μέτρα θα είχαν προληφθεί αυτές οι επιθέσεις. Η αστυνομία ήταν εκεί. Γιατί δεν μπόρεσαν να αλλάξουν την κατάσταση. Γιατί ίσως δεν τολμήσαν να σταματήσουν αυτά τα γεγονότα. Δεν νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά είναι αποδεκτά και δεν μπορούμε να παραμείνουμε σιωπηλοί. Ευχαριστώ. Opinia publică românească, precum și presa din România. Κύριε Τανσίλα, ε, στην Ρουμανία τα μαζικής ενημέρωσης ε, ε, μιλούν για την οικογένεια Μποντνάρη, ε, της τα παιδιά συνελήφθησαν στην Νορβηγία. Οι νορβηγικές αρχές, δεν ξέρουμε γιατί οι νορβηγικές αρχές πήραν αυτή την απόφαση. Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση. Η έλλειψη πληροφοριών είναι αποτέλεσμα της έλλειψης διαφάνειας από πλευράς των νορβηγικών αρχών. Η Νορβηγία προφανώς δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ο πατέρας αυτών των παιδιών ε, είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστεύω ότι είναι σημαντικό ο ίδιος και η οικογένειά του να τύχουν προστασίας από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Οι ρουμανικές αρχέ δεν κάνουν όμω κάτι τέτοιο προ το παρόν. Θα ήθελα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στηρίξει την, το αίτημά μας ε, οι εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων να εμπλακούν ενεργά για να διευκρινιστεί η κατάσταση των πέντε παιδιών της οικογένειας Μπονταρίου. Η κυρία Φωτίγκα. Ευχαριστώ. Δύο ε, ευρωπαϊκοί καθισμικά όργανα ε, αποφάσισαν να ελέγξουν ε, την χώρα μου, την Πολωνία, για την εφαρμογή των κανόνων Πρόκειται για το παράγωγο δίκαιο ε, που τίθεται σε εφαρμογή εδώ με τρόπο κατασταλτικό και εφαρμόζει και διπλά μέτρα και σταθμά απέναντι σε κάποια νέα κράτη-μέλη και στο έθνη τους, όπως και απέναντι και σε διαφορετικές ε, ε, κυβερνητικές υπηρεσίες όπου χειρίζεται τα θέματα αυτά. Ο κύριος Τζάκοφτσιτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η δημιουργία των φρακτών με ασυρματόπλεγμα μεταξύ Σλοβενίας και Κροατίας έχουν δημιουργήσει μεγάλη αναταραχή στους πολίτες και των δύο χωρών. Οι διαδηλωτές, οι διαμαρτυρώμενοι διαδηλωτές παίξανε βόλεϊ πάνω από αυτό το φράκτη. Ο φράκτης αυτός δημιουργήθηκε σε περιοχές όπου κανείς δεν μπορούσε να περιμένει μαζική είσοδο μεταναστών. Αυτό ήταν λοιπόν μια ανεύθυνη ενέργεια και κατά των Κροατών και κατά των Σλοβαίνων και κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι φράκτες αυτή με συνέχεια είναι μεγάλος κίνδυνος για τους κατοίκους των περιοχών αυτών και γι' αυτό το λόγο θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητήσει αμέσως την καταστροφή αυτού του φράκτη με σειρματόπλεγμα μεταξύ των δύο χωρών μας γιατί είναι μια άμεση απειλή στην ασφάλεια των πολιτών μας. Ευχαριστώ. Ο κ. Φερέιρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, πολύ προπαγανδίζεται η Τραπεζική Ένωση, αλλά αυτό που βλέπουμε στην Πορτογαλία είναι ακόμα τραπεζικό σκάνδαλο που ε, δείχνει την αδυναμία του συστήματος εποπτείας ε, είναι μια απάτη αυτή η Τραπεζική Ένωση και το σύστημα εποπτείας. Ε, ένα δισεκατομμύρια ευρώ δόθηκαν στην Μπανίφ το 2013 και τώρα στην πράξη τι συμβαίνει. Το πορτογαλικό κράτος χρηματοδοτεί 2,5 με 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ μια ξένη ευρωπαϊκή τράπεζα για να εξαγοράσει την Πανίφ και να μπει στην εθνική αγορά. Δηλαδή το κράτος ε, θέλει να πληρώσει τα χρέη της τράπεζας Μπανίφ ε, έτσι ώστε να δοθεί καθαρή και αγνή χωρίς χρέη στη Ισπανική τράπεζα, στην Πάγκο Σανταντέρ. Όλα αυτά α, ε, δείχνουν τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. θα υποβάλουμε και γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζουμε θα την απαντήσει σύντομα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η απάτη της Volkswagen όπου ε, έχει <clears throat> παρα, παραποιήσει τα στοιχεία πολλών αυτοκίνητων, εκατομμυρίων αυτοκίνητων για να, χιλιάδων αυτοκίνητων για να κρύψει τις εκπομπές τους, αυτό είναι μια πραγματική απάτη για τους καταναλωτές που θέλουν να αγοράσουν υποδειγματικά καθαρά αυτοκίνητα. Είναι απάτη για τις δημόσιες αρχές. Μόνο στην Ισπανία πουλήθηκαν 50.000 από αυτά τα ε, μαγειρεμένα αυτοκίνητα τα οποία είχαν απαλλαγή από πολλούς φόρους. Ακόμα δεν ξέρουμε πόσα χρήματα έχει χάσει από αυτό η δημόσια αλλά είναι πολλά εκατομμύρια. Στη Ναβάρα και στην Καταλωνία <clears throat> η Volkswagen πήρε 300 εκατομμύρια άμεσες κρατικές επιδοτήσεις. Πάρα πολλοί πολίτες έχουν υπό υποφέρει λόγω μια επιχείρηση η οποία έκανε τέτοιε απάτε. Θα πρέπει η Επιτροπή Έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αναλύσει τα γεγονότα και να ζητήσει απόδοση ευθυνών. Δεν μπορεί λοιπόν να γίνει κάτι άλλο γιατί αυτή τη στιγμή διακυβεύεται η ίδια η έννοια τη υπηκότητά μα. Ευχαριστώ κύριο Μάτ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες ε, και κύριοι, όταν η τσεχική δημοκρατία μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλοί συμπατριώτες μου θεωρούσαν ότι η ένταξη θα μειώσει τη διαφθορά, θα ενισχύσει τη δημοκρατία στη χώρα και θα φέρει ευημερία. Σήμερα όλοι βλέπουν ότι αυτές ήταν φρούδες ελπίδες που καταρακώθηκαν. Όλοι στη Τσεχική Δημοκρατία βλέπουν ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια αύξησαν τη διαφθορά. Ε, εν ώψη της προσφυγικής ε, κρίσης φάνηκε η αντιδημοκρατική φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απομονώθηκε από τον τσεχικό λαό. Εις επίμετρον βλέπουμε σήμερα ότι ε, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει παραγνωριστεί ε, με το πρόσχημα ότι είναι κατεπήγοντα τα θέματα. Οι περισσότεροι πολίτες στο Ευρωπαϊκό, στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι υπέρ του Brexit και αυτό δεν με εκπλήσει βέβαια. Ευχαριστώ κύριος Μποργκέτσιο. Ευχαριστώ. Στην Ιταλία έχουμε το σκάνδαλο της χρεοκοπίας τεσσάρων τοπικών επιχειρήσεων και έχουμε ζητήσει ήδη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιληφθεί. Θέλω να επιστήσω την προσοχή του, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ανάγκη να πιέσει την κυβέρνηση της Ιταλικής κυβέρνησης να αποζημιώσει τα θύματα αυτών των επιχειρήσεων. Γιατί όλοι αυτοί οι ομολογιούχοι οι οποίοι ε, επένδυσαν όλες τις αποταμιεύσεις τους ήταν άτομα τα οποία πολλές φορές είχαν τραγικό τέλος. Ένας ε, από αυτούς αυτοκτόνησε πρόσφατα. Υπάρχουν πολλοί λοιπόν μικροί καταθέτες οι οποίοι πρέπει να αποζημιωθούν 100% γιατί πραγματικά τους κορόιδεψαν με το να τους πουλήσουν τίτλους οι οποίοι δεν είχαν καμία εγγύηση όπως είχε παρουσιαστεί από το προσωπικό της τράπεζας και είχαν αποκρύψει απόλυτα την πραγματικότητα η οποία τώρα έχει έλθει στην ε, επιφάνεια με την τράπεζα της Ετρουρίας που είναι μία από αυτές επίσης τις τράπεζες. Θα πρέπει λοιπόν ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου να λάβει υπόψη αυτή την ε, αναφορά και να ε, αποτίσει και φόρο τιμή στο πρώτο θύμα αυτής της απάτης που έχασε στη ζωή του. Κύριος Ζαριανόπουλος. Μάικρο, στην ελλάδα η κυβέρνηση σύριζα ανέλ αναλαμβάνοντα τη βρώμικη δουλειά υλοποιώντα μνημόνια και ευρωνοσιακέ συνθήκε ικανοποιεί την απέτηση του κεφαλαίου για παραπέρα κατεδάφιση κοινωνική ασφάλιση απαλλαγή τη εργοδοσία και του κράτου από την ευθύνη του ακόμα φθηνότερη εργατική δύναμη εξοικονόμηση δισεκατομμυρίων ενίσχυση στο κεφάλαιο. κανεί δεν ξεφεύγει. παλιοί και νέοι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι αγρότε αυτοαπασχολούμενοι γυναίκε ιδιαίτερα οι νέοι που λόγω περιπλάνησης μεταξύ ανεργίας και ελαστικών σχέσεων εργασίας θα αρκεστούν όπως η συντριπτική πλειοψηφία σε σύνταξη επίδομα πείνας σε περασμένη ηλικία. ενώ επικαλείται τη βιωσιμότητα άδειων ασφαλιστικών ταμείων που κατάκλεψαν όλες οι κυβερνήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων στέλνει νέους πελάτες σε ιδιωτικές ασφαλιστικές και με την οδηγία solvency ii τις ενισχύει με κεφάλαια για να ξεκοκαλιστούν πάλι ασφαλιστικά αποθεματικά σε επενδύσεις επιχειρήσεων και χρηματιστήρια η κυβέρνηση αποζητά και για το μνημόνιό της δημοκρατική νομιμοποίηση του εγκλήματός της από το ευρωκοινοβούλιο αποκαλύπτοντας τον αντιδραστικό ρόλο του. ο λαός αρνείται την σφαγή της κυβέρνησης οργανώνεται παλεύει με διαδηλώσεις γενικές απεργίες για να μην φτάσει το αντιασφαλιστικό έκτρωμα στη βουλή. Ε, Ευχαριστώ η φορολογική μας ε, πολιτική επηρεάζει και το περιβάλλον για τη δημιουργία θέσεων επασχόλησης. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι η κυριαρχικότητα στο φορολογικό τομέα και η ε, φορολογική, φορολογικός ανταγωνισμός μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτό το οποίο βλέπουμε, αλλά θα μπορούσαμε να κάνουμε με κάποια μεγαλύτερη εναρμόνιση πολύ περισσότερο για να έχουμε πιο κοντινές ε, τιμέ για το ΦΠΑ, συντελεστέ ΦΠΑ. Αυτό δεν θα βοηθήσει μόνο το ηλεκτρονικό εμπόριο, θα βοηθήσει και τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Θα πρέπει επίση να υποστηρίξουμε αυτέ τι επιχειρήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τη βελτίωση τη διαχείριση των κανόνων και να εξασφαλίσουμε λοιπόν τη συμπλήρωση εσωτερική αγορά. Νομίζω ότι η ενιαία <clears throat> καταγραφή ΦΑΠ και ε, η, μόνη, η μία μονάχα καταγραφή για κάθε εταιρεία θα βελτιώσει την κατάσταση των μικρών επιχειρήσεων και θα δημιουργήσει και πολλές νέες επιχειρήσεις και έτσι οι πολίτες μας θα έχουν πολλαπλά ωφέλη. Κύριε Καρτίνη. Κύριε Πρόεδρε, στη χώρα μου η οικογένεια είναι πολύ σημαντική και κατά παράδοση παιδιά και γονείς παραμένουν ενωμένοι στην οικογένεια. Μια πρόσφατη μελέτη που έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο δείχνει ότι η Ρουμανία είναι η χώρα όπου είναι τα πιο ευτυχισμένα παιδιά. Η περίπτωση της οικογένειας Μποντναρίου και όχι μόνο έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο λόγω του πώς χώρισαν οι νορβηγικές αρχές τα παιδιά από τους γονείς που δεν ήθελαν. Οι διαδικασίες δεν ολοκληρώθηκαν. Τα δικαιώματα των παιδιών ρυθμίζονται στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το συμφέρον του παιδιού πάντοτε είναι το σημαντικότερο. Η Νορβηγία έχει προσυπογράψει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Παιδιών και αναρωτιέμαι τι κάνουμε για να υπερασπιστούμε τους πολίτες μας που ζουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης η, Ευρωπα... η Ευρώπη, το Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν να παρέμβουν ούτω ώστε να επανενωθεί η οικογένεια αυτή. Μητέρα είμαι και εγώ και δεν νομίζω ότι κανείς θα μπορούσε να αγαπήσει τα παιδιά περισσότερο από τους φυσικούς γονείς τους. Αύριο την 3η 19 ξεκινάει ε, η Ισπανία η δίκη εναντίον του Ρόλ Καπίν, ε, φωτογράφου. Ε, πρόκειται για μια ποινικοποίηση, μια δίωξη, πολιτική δίωξη του Ισπανικού κράτους εναντίον μέσω μαζικής ενημερώσεις που επικρίνουν την κυβέρνηση. Ε, το ίδιο βλέπουμε ε, και με άλλους ακτιβιστές. πρόκειται για επίθεση εναντίον της ελευθερίας του τύπου και κάτι που προστίθεται στις στις, ε, σε άλλες ε, δράσεις εναντίον της ελευθερίας του λόγου ε, και υπέρ της λογοκρισίας. Είναι φαινόμενα συχνά τα τελευταία χρόνια στην Ισπανία και λαμβάνουν χώρα εναντίον αυτών που αντιδρούν όπως ο Ραούλ Καπίν που δημοσιεύοντας φωτογραφίες όπως αυτές. Γιατί ότι δεν είναι έγκλημα η ενημέρωση. Απαιτούμε το τέλος της καταπίεσης και των διώξεων εναντίον αυτών που την καταγγέλνουν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σόλτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να απαντήσω στον κύριο Γιακότσης. Δεν μου αρέσει δεν μ' αρέσει το αγκαθωτό σύρμα, το κοφτερό αγκαθωτό σύρμα στα σύνορα. Έχω δει και ο ίδιος πως μεγάλη ζημιά μπορεί να κάνει αυτό το ε, σύρμα σε αυτούς που ζουν στην περιοχή και στα ζώα που ζουν εκεί. Η Σλοβενία δεν δημιούργησε αυτό το φράκτη επειδή της άρεσε. Έπρεπε να το κάνει για να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά υπάρχει κίνδυνος να υπάρξει φαινόμενο ντόμινο. ο Υπουργό Εξωτερικών της Κροατίας είπε ότι αυτό μπορεί να επαναληφθεί σε άλλες χώρες των Βαλκανίων. Γιατί οι μετανάστες αλλάζουν τις διαδρομές. Ο κ. Μπάτεν. Ευχαριστώ. Πολλοί από τους εκλογείς μου έχουν αναφερθεί στην οδηγία για τα πυροβόλα όπλα, ιδίως από το Αυτοκρατορικό Μουσείο, το Μουσείο Πολέμου και τα Βασιλικά ε, Οπλοστάσια. Δεν θέλουν να καταστραφούν οι ιστορικές αυτές συλλογές και να μην μπορούν να πάρουν περισσότερα όπλα. Αυτή η τροπολογία είναι μια πανικόβλητη αντίδραση στις, στα γεγονότα του Παρισιού. Πόσες τρομοκρατικές ενέργειες έχουν γίνει με ε, όπλα αντίκες. Καμία βέβαια. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν μια εξαίρεση για τα μουσεία και αυτή θα πρέπει να ισχύει για όλους αυτούς που, αγορά, που αγοράσουν ή συλλέγουν όπλα αντίκες. Θα πρέπει οι βουλευτές να το υποστηρίξουν. Και αυτό είναι το τελευταίο παράδειγμα του ενδιαφέροντος των εκλογέων μου που θίγεται από ανόητη και όχι σωστά σταθμισμένη νομοθεσία. Εγώ θα τους έλεγα να πάρουν τα όπλα, μεταφορικά φυσικά, και να αγοριστούν για την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο επερχόμενο δημοψήφισμα. Merci, Monsieur le ο κ. Λεμπρετών, η Κομισιόν ξεκίνησε μια έρευνα εναντίον διαφόρων συνδικάτων ε, Γάλλων Γεωργών ε, γιατί υποτίθεται ότι παραβίασαν το άρθρο 101 της Συνθήκης της Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, του ανταγωνισμού και ενδεχομένως ε, θα τους επιβληθούν σημαντικά πρόστιμα. Αυτή η πρωτοβουλία της Κομισιόν από οικονομικής ε, πλευράς είναι υπερβολική και σκανδαλώδης από ανθρωπιστικής πλευράς. Στη Γαλλία χιλιάδες ε, κτηνοτρόφοι και παραγωγή γάλακτος ε, πεθαίνουν από τις καταστροφικές αποφάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το τέλος των ποσοστώσεων, το ρωσικό εμπάργο ε, και ε, οι, ε, ε, οι χιλιάδες Αζερβαϊτζανοί, οι οποίοι έχουν προσληφθεί από τους Γερμανούς, έχουν δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην, στους Γάλλους κτηνοτρόφους. Είναι απαράδεκτο η Κομισιόν σήμερα να τους κατηγορεί. Ε, η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση ε, θα βρει απέναντί της το γαλλικό λαό. Στην Βρετάνια έχει ήδη ξεκινήσει ο ξεσηκωμός. Ξεσηκωμός αν όχι και επανάσταση. Ο κύριος Ρολάν, ο πρόεδρος της Επιτροπής <clears throat> έχει καταγγείλει εδώ την ύπαρξη ενός 29ου κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, έθνους που απαρτίζεται από τους άνεργους. Δεν μπορούμε να δεχτούμε 7 εκατομμύρια νέων να είναι χωρίς εργασία και χωρίς κατάρτιση. Δεν μπορούμε να έχουμε πάνω από 10% των νέων που αποχωρούν πρόωρα από το σχολείο. Υπάρχουν συστήματα που διευκολύνουν τη μετάβαση μεταξύ σχολείου και απασχόλησης. Έχουν λειτουργήσει στα κράτη-μέλη μας. Η εναλλασσόμενη παιδεία, κατάρτιση είναι κάτι το οποίο έχει λειτουργήσει και έχει βοηθήσει και τους κοινωνικούς εταίρους. Επίσης το έρασμος είναι μια μεγάλη επιτυχία για κατάρτιση, για κινητικότητα. Ο έρασμος είναι ένα πολύ σημαντικό εκολαπτήριο Ευρωπαίων εργαζομένων. Ας χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να αντιμετωπίσουμε την ανεργία των νέων με ένα πραγματικό σύστημα ε, εναλλασσόμενης κατάρτισης και μαθητείας για τους νέους. Όταν υπάρχουν λύσεις έχουμε την υποχρέωση να τις εφαρμόσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Παπαρδέλ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, αναφέρομαι στην περίπτωση αυτή στην Ορβηγία, όπου αποχωρίστηκαν ε, τα παιδιά από τους γονείς. Ε, στη Νορβηγία το 2014. Ε, υπάρχουν και άλλες τέτοιε περιπτώσεις. Πόσα είναι αυτά τα παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οικογένεια Μπορναρίου έχασε τα πέντε παιδιά της ε, για λόγους που δεν αιτιολογήθηκαν σωστά από τις νορβηγικές αρχές χωρίς εντολή του δικαστηρίου, χωρίς σωστή λήψη αποφάσεων, χωρίς να, δοθούν, ε, να δοθεί τεκμήριο αθεότητα στην οικογένεια. Και δεν είναι μόνο αυτή η περίπτωση. Δείχνει την, τον τρόπο που λειτουργούν οι νορβηγικές αρχές γενικότερα. Θέλω να ζητήσω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεννοηθούν ε, με τους ε, ομολόγους τους για να διασφαλιστούν τα δικαιώματα της οικογένειας. Ε, αυτό προβλέπεται άλλωστε και από το νόμο για την ηθαγένεια. Θα πρέπει οι πολίτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προστατευτούν απέναντι σε τέτοιου κινδύνου. Ο κύριος Κάρβερ. Η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μέση Ανατολή αμφισβητείται και πάλι και η νομοποίησή της. Ε, μια μη κυβερνητική οργάνωση ε, ε της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, υποστηρίζει τους ε, Παλαιστινίους ε, δήθεν και τους όμως δημιουργεί μια στην παγίδα έτσι ώστε να πουλήσουν τις, τις περιουσίες τους στους Ισραηλινούς. Αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση παίρνει λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι παράδειγμα Τον περασμένο μήνα πήρε 30.000 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Δημοκρατία. Ο Έλμαρ Μπρόκ είναι στο δικό Συμβούλιο του Ταμείου αυτού, μαζί με άλλους εννέα ε, ευρωβουλευτές. Ε, κύριε Πρόεδρε, επί τη ευκαιρία, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, αίμα στα χέρια της. Ευχαριστώ. Κύριος Μπούντα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα θεσμικά όργανα πρέπει να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούν να παρακολουθούν απαθώς βλέποντας τη δράση των νορβηγικών ε, υπηρεσιών που καταστρέφουν τις οικογένειες ε, ε, θεωρείται ότι η πίστη στο Θεό ε, πρέπει να τιμωρηθεί. Παίρνουν τα παιδιά ε, από τους γονείς. Αυτή είναι η περίπτωση Μποντναρίου που έχασε τα πέντε παιδιά τους και το πιο μικρό θυλάζει ακόμα γιατί είναι τριών μηνών. Είναι, αυτό επηρέασε πολύ την ανάπτυξή τους. Τρεις χιλιάδες παιδιά σήμερα είναι τα θύματα δικαστικών αγώνων μεταξύ των γονέων για την επιμέλεια. Αλλά Κανείς ε, δεν μπορεί να μην αιτιολογεί επαρκώς την ε, απόφαση αποχωρισμού των παιδιών από τους γονείς. Ε, ελπίζω να αναθεωρηθεί η πολιτική σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ κύριε Φερνάνδης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να επιστήσω την προσοχή των βουλευτών στις τρομερές πυρκαγιές που έπληξαν τη Βόρεια Ισπανία το Δεκέμβριο και ιδίως στην περιοχή των Αστούριας πάνω από 453 εστίες ε, πυρός, οι περισσότεροι εμπρισμοί στη νύχτα 29 με 30 ε, Δεκεμβρίου 2015, από τις οποίες το 1 τρίτο στην περιοχή του Αστούριας, που είχαν μεγάλο αποτέλεσμα στο σύνολο της περιοχής. Εγώ είδα επιτοπίως ποια ήταν η κατάσταση και το τελικό αποτέλεσμα αυτών των ε, ε πυρκαγιών. Όλη η περιοχή λοιπόν των Αστούριας ήταν το θύμα πάνω από 100 πυρκαγιών που ήταν ένα μεγάλο μέρος εμπρισμοί. Η κυβέρνηση των Αστούριας προσπαθεί να βρει τρόπο για να αποζημιώσει τα άτομα, τα νοικοκυριά που καταστράφηκε το σπίτι τους, τα χωράφια τους, τα ζώα τους και είναι απαραίτητη η κυβέρνηση να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει τα απαραίτητα. Εγώ ζητώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βοηθήσει ώστε να μπορέσει να καταπραίνει λιγάκι τα αποτελέσματα αυτών των τρομερών πυρκαγιών στην Αστούρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Τόμοκ. Η κυρία Τόμοκ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως η ε, κυρία Γκάλ Πέλτς, θα ήθελα και εγώ να μιλήσω για την ε, ε, βία της οποίας είμαστε μάρτυρες στην Ευρώπη τελευταία. Δεν υπάρχει καμία αποδεκτή εξήγηση, καμία δικαιολογία. Ορισμένα, σε ορισμένα φόρουμ βέβαια κάποιοι δείχνουν να επιχαίρουν για τη βία αυτή εναντίον των γυναικών. Χρειάζονται, χρειάζεται η, προφανώς να εκπαιδευτούν οι πρόσφυγες, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Χρειάζεται μια συνολική αντιμετώπιση της ένταξής τους. Αυτοί που έρχονται στις πατρίδες μας θα πρέπει να βοηθηθούν, θα πρέπει να στηριχθούν, αλλά ταυτόχρονα αναμένουμε από αυτούς ότι θα σέβονται την, το, την κουλτούρα μας, τα έθιμά μας, τα ήθη μας και ότι δεν θα προβαίνουν σε πράξεις βίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούσατε τους συναδέλφους. Εκπροσωπούμε την κοινή γνώμη στη Ρουμανία που ε, έχει εντυπωσιαστεί από την ε, αφαίρεση των παιδιών από την οικογένεια Μποτναρίου από τις κοινωνικές υπηρεσίες της Νορβηγίας ε, χωρίς καμία απόφαση δικαστηρίου μέσω μιας ε, δυσανάλογης ε, ε πράξης ε, κατά παράβαση των διεθνών συνθηκών περιπροστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού. Ε, οι νορβηγικές αρχές έχουν ήδη καταδικαστεί για προηγούμενη τέτοια περίπτωση ε, από το ε, Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ελπίζω ότι όλοι μας θα κινητοποιηθούμε και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ίδιο έτσι ώστε να πιστούν οι νορβηγικές αρχές να βελτιώσουν το νομοθετικό τους πλαίσιο έτσι ώστε να μην επαναληφθούν τέτοιου είδου φαινόμενα. Κύριος Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Οι Ισπανικές αρχές αποφάσισαν μονομερός πριν από λίγες μέρες να θίξουν πάνω από 500 είδη πτηνών και περίπου 500.000 άτομα που ζουν στο δέλτα του Εύρου. Τα σχέδια υδρολογικού χαρακτήρα έχουν επικριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχουν αναφέρει ιδιαίτερα τις παραλήψεις και τα ασφάλματα των Ισπανικών αρχών για την οδηγία για τα σχέδια ε, περί λεκανών, ε, υδροροϊκών λεκανών. Είναι απαραίτητο λοιπόν να τονίσουμε ότι η προστασία των περιοχών δεν εξασφαλίζεται από τα σχέδια αυτά και εξακολουθούν και τα νέα σχέδια να έχουν το ίδιο πρόβλημα. Θα πρέπει η Κομισιόν να δράσει αμέσω και να επαναφέρει αυτά τα προγράμματα στι Ισπανικέ Αρχέ για να τα αλλάξουν. Υπάρχει κίνδυνο <coughs> για τη διατήρηση όχι μόνο ενό συστήματο αλλά και για την επιβίωση χιλιάδων Ευρωπαίων πολιτών. Πρέπει λοιπόν να δράσουμε τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και ο πρόεδρος. Κυρία Σαμπόρσκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Θέλω να εκφράσω αλληλεγγύη με τις γυναίκες που έζησαν τη βία, την παρανόχληση, τις απειλές στην κολονία της Γερμανίας. Δεν ανεχόμεθα τέτοιες συμπεριφορές στην Ευρώπη. Είμαστε υποχρεωμένοι να, υπο... να υπερασπιστούμε την αξιοπρέπεια κάθε γυναίκας. Δεν έχει σημασία αν οι... αυτοί που έκαναν την επίθεση ήταν πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μετανάστες. Το σημαντικό είναι ότι είναι απαράδεκτη η συμπεριφορά. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε δίπλα μέτρα και σταθμά όταν κρίνουμε τέτοια ε, αδικήματα. Τα συμβάντα στην κολονία δείχνουν ότι αντιμετωπίζουμε μεγάλες προκλήσεις. Ας τις πάρουμε στα σοβαρά, χωρίς όμως ε, να κάνουμε επιφανειακές ε, κρίσεις Ευχαριστώ πολύ και τελειώνει το τμήμα αυτό τη συζήτηση. Αύριο το πρωί στι 9 είναι η επόμενη συνεδρίασή μα από τι 9 τι 14.30 και από τι 15 τι 23. Η μέση διάταξη τη αυριανή μέρα έχει δημοσιευτεί και είναι στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κλείνουμε τη συνεδρίαση. Ευχαριστώ τους ε, διερμηνείς οι οποίοι και πάλι με υποδειγματικό τρόπο